Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ, καθίστε. Ξεκινάμε το ψήφισμα το οποίο αφορά την ελευθερία έκφραση στο Βιετνάμ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο ψήφισμα για την Καμπότζη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε Έχασα την παράγραφο 12. Παράγραφος 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα για το Ελσαλβαδόρ. Έχουμε πρώτα μία πρόταση ψηφίσματος δύο ομάδων σε ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο κοινό ψήφισμα τεσσάρων ομάδων. και έχουμε... Έχει ζητήσει τον λόγο η κυρία Σκοτ Κέιτο. Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω μία προφορική τροπολογία σε σχέση με κάτι το οποίο συνέβη χτες το βράδυ. Πρέπει να αλλάξουμε το εκτιμώντας γάμο στο τέλος να λέει ενώ αφού πέρασε τα τελευταία δέκα χρόνια στην φυλακή η Τεοδόρα Βάσκες εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό 13 Δεκεμβρίου 2017 και απορρίφθηκε η αίτησή της, η έφεσή της. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για αυτήν την προφορική τροπολογία. Όχι. Οπότε θα ψηφίσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή το ψήφισμα στο σύνολό του, όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Περνάμε τώρα στην έκθεση Κουτιέρες. Ψηφίζουμε το ψήφισμα της Επιτροπής ε, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ντάντι για να μιλήσει εξ ονόματος ε, της Αρμόδιας Επιτροπής. Έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εξ ονόματος του εισηγητή Σέρτζο Γκουτιέρες, καλώ το σώμα να υποστηρίξει την έντολη ε, που προκύπτει ύστερα από διαπραγμάτευση και που εγκρίθηκε την προηγούμενη φορά από την, την προηγούμενη εβδομάδα από την Επιτροπή Αγοράς για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μέσα στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Πρέπει να υποστηριχθεί η τροποποίηση στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να γίνει σεβαστή η δημοκρατική νομιμότητα των τοπικών συνελεύσεων και εθνικών κοινοβουλίων. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ευρύτατη πλειοψηφία που εξασφαλίστηκε στην ψηφοφορία στην Επιτροπή θα επιτρέψει και στον εισηγητή να ξεκινήσει τον τριμερή διάλογο με ισχυρή και σαφή εντολή. Γι' αυτό εκ μέρους του εισηγητού σας καλώ να υποστηρίξετε την εντολή του για διαπραγμάτευση. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Ντέντη. Ντάντι, θέλει κανείς να, σταθεί, να στραφεί κατά της πρότασης. Κύριος Ντεϊόγκ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ομολογώ ότι προσπάθησε το Κοινοβούλιο να βελτιώσει την κακή πρόταση της ε, Κομισιόν, αλλά ε, παρόλα αυτά πρόκειται για μια αναβολή των ε, εθνικών δημοκρατικών αποφάσεων για τρεις με έξι μήνες. Και οπωσδήποτε αυτό έχει αντίκτυπο στο πώς φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά δηλαδή το ότι θα πρέπει να ε, εκφραστεί πρώτα η Κομισιόν πριν σχηματιστούν ε, τοπικά συμβουλία. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Jong. Περνούμε στην ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψήφισμα για την κατάσταση στο Αφγανιστάν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματος για την κατάσταση της μειονότητας στο Ροχίνγκια. Παράγραφος 4. Πρώτη τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 στο αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε είπε κατά αποχές εγκρίνεται έκθεση Κοράτσα Πίλτ η συγκήτρια για ένα λεπτό Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τους συναδέλφους για την θερμή υποστήριξή τους. Ας προσπαθήσουμε σήμερα να στείλουμε ένα ηχηρό ε, και ισχυρό μήνυμα προς τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να δράσουν ε, ταχύτερα και να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν τα παιδιά και από κοινού με την κοινωνία των πολιτών, ε, την, τον κλάδο IT, τις αρχές επιβολής του, νόμου, να έχουμε μηδενική ανοχή στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών on και offline. Θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στα έργα και να παραμείνει η Ευρώπη ένας ασφαλής χώρος για όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, και ψηφίζουμε. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχέ απερίφθη, 2 υπέρ κατά αποχέ απερίφθη, 3 σε δύο τμήματα, το πρώτο παρακαλώ υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, δεύτερο υπέρ, κατά αποχέ απερίφθη, 4 υπέρ, κατά αποχέ απερίφθη, τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση άρχεται ψήφισαν όλοι πέρασε Εγκρίνεται. Έκθεση Μαριά. Τροπολογία 3-2 τμήματα. Το Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Παράγραφος 4 αρχικό κείμενο υπέρ. Επαληθεύουμε το 3 στο δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία παρακαλώ. Τροπολογία 3 δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Παράγραφος 4 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 5 του αρχικού κειμένου, δύο τμήματα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος τροπολογία 4 ονομαστικά άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και απερίφθη. Τροπολογία 18, ονομαστική εκκλησία, άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 5 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη, αρχικό κείμενο στην Παραφή 22, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Επαληθεύουμε, άρχεται η ψηφοφορία, δεύτερο τμήμα του αρχικού κειμένου της παραγράφου 22. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6, ονομαστική κλίση, άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7, δύο τμήματα. Το πρώτο, ονομαστικά, άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστικά. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 11 ονομαστικά. Άρχεται. Ψήφισαν όλα. Πέρας. Απερίφθη. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 17 ονομαστικά άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. Τροπολογία 1, σε δείχνει με τα πρώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ε, τροπολογία 14 ονομαστικά άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Την τροπολογία 10 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται λογική σκέψη Ο, αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. λογική σκέψη ΤΑΦ T, αρχικό τμήμα πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ, Επαληθεύουμε το, την τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη και στο συγγνώμη. Δεύτερο, ε, τροπολογία 2 υπέρ κατά. Εγκρίνεται 16. Εντάξει, αλλά ήταν τα ίδια ποσοστά. Ε, τη 2. Άρχεται, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Eichhout. 18 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 αρχικό κείμενο. Δύο τμήματα πρώτο. Ονομαστικά κάθε φορά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Ε, τις Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 2. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. Αρχική παράγραφος 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε παρακαλώ, άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 45 του αρχικού κειμένου. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 46 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με τις ίδιες πλειοψηφίες 81 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 85, δύο τμήματα, ονομαστικά κάθε φορά. Το πρώτο παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται δεύτερο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και περίφθη. Ονομαστική κλίση στην παράγραφο 86 αρχικό κείμενο άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 89 υπέρ κατά. Είναι πολύ στενές οι πλειοψηφίες σας, θα επαληθεύσουμε λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 93 ονομαστική Εκκλήση Άρχεται», Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 113 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Όχι, ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το ψήφισμα στο σύνολό του όπω τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας και εγκρίθηκε. Και υπενθυμίζω ότι σημειώνεται η, η ψήφο σας ε, όταν ε, αφαιρέσετε την κάρτα από το μηχάνημα. Σας εύχομαι καλή επάνωδο. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα συναντηθούμε στις Βρυξέλλες. Σας εύχομαι Καλό Πάσχα, χρόνια πολλά στο Αρμίς. Ευχαριστούμε πολύ και τις υπηρεσίες, λέει ο Πρόεδρος. Και όποιος είναι εδώ για τις επεξηγήσεις ψήφου, παρακαλώ να ετοιμαστεί να λάβει το λόγο. Όποιος δεν θέλει να παρακολουθήσει επεξηγήσεις ψήφου, να αποχωρήσει πάρα χρήμα. οπωσδήποτε οι διάδρομοι προσφερόνται πολύ περισσότερο για αγκαλιές, φιλιά και αποχαιρετισμούς για τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό παρακαλώ να επιτραπούν αμφότερες δραστηριότητες με ηρεμία. Und Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου να σημειώσουμε πρώτα στα πρακτικά ότι ευχήθηκα κατά λάθο καλό Πάσχα, προφανώς εννοούσα καλά Χριστούγεννα.